good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. Unfortunately, it's coming to an end. And... Καλημέρα σε όλους. Ε, ξεκινάει η σημερινή συνεδρίαση. Σήμερα, λοιπόν, ε, βλέπω ότι είσαστε όλοι εδώ, με μεγάλη μου χαρά. Κάποιοι, όπως ο Ματίας, ε, λείπουν ακόμα σε διακοπές. Θα μας έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Καταρχάς λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι. Έγκριση των πρακτικών της ε, συνεδρίασης τη 11 η Ιουλίου. Ε, αν υπάρχουν παρατηρήσει, στείλτε ε, στο γραμματέα. Πάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταρχάς να σας πω ότι έχουν αλλαγές στο Συμβούλιο ε, του SRB, του ε, Συμβουλίου, Ενιαίου Συμβουλίου ε, και ο κύριος Γκένινγκ ε, μας ενημέρωσε ότι θα φύγει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόλις βρεθεί διάδοχος. Επίσης η Κομισιόν ανέφερε μια, στην ε, επίσημη εφημερίδα ότι η Επιτροπή θα εμπλακεί στην επιλογή των ε, συντονιστών. Σύντομα θα ε, έχουμε νέα για αυτή τη διαδικασία. Με την ευκαιρία να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω την κυρία Κέλερμαν. Επίσης, διοργανικές διαπραγματεύσεις Έχουμε τον ε, τριμερή διάλογο για, την, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 849 του 2015 είναι η οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα επόμενα σημεία συζητήσεων συζητήθηκαν. Έχουμε την εθνική και περεθνική αξιολόγηση κινδύνων για την ενιαία εποπτική αρχή ε, ασφάλεια ζωής, αποκάλυψη πληροφοριών, υποχρέωση των επιτροπών να ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εθνικές νομοθεσίες και τις κυρώσεις. Φαίνεται ότι ο διάλογος έγινε με επικοδομητικό πνεύμα. Από όλες τις πλευρές όμως επί της ουσίας δεν έγινε πρόοδος. Ε, δεν υπήρξε πρόοδο. Καλή διάθεση, αλλά καθόλου αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Η Προεδρία θα κάνει δύο ε, ομάδες εργασίας ε, το Σεπτέμβρη για να προετοιμάσει τον επόμενο πολιτικό τριμερή διάλογο που είναι στις 3 Οκτωβρίου τις γερμανικές, δηλαδή διακοπές την αργία στη Γερμανία στο Στρασβούργο και ελπίζουμε ότι τότε θα υπάρχει πρόοδος, γιατί για μας το EMLD5 είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στο σημείο 5 στα μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που δρούν για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ε, έχουμε η συγγήτρια, την κυρία Μόρις Σκοτ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να καλωσορίσω τους βουλευτές που τα κατάφεραν να έρθουν εδώ. Είναι εντυπωσιακό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα είχαμε μία συνάντηση των σχεδόν λίγο πριν τις διακοπές. Πήγε πολύ καλά, υπήρχε καλό πνεύμα συνεργασίας, καλή διάθεση, μεγάλη πρόοδος, μεγάλη σύμπνοια μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Θα έχουμε άλλη μία συνάντηση των σχεδόν σήμερα το απόγευμα και αδειμονώ και τότε να έχουμε μία καλή συνάντηση. Οι καταγγέλτες παίζουν σημαντικό ρόλο για το δημόσιο συμφέρον, όπως ξέρετε. Παρά όμως ε, τα πιθανά ωφέλη, μόλις έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει νομοθεσία για την προστασία τους. Από τις έξι αυτές ε, ε, χώρες, όλες, επέλεξαν οριζόντια προσέγγιση. Η ομάδα μου, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και εδώ, θεωρούν ότι η προστασία πρέπει να επεκταθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι καταγγέλτες θα πρέπει να, υπο... να προστατεύονται σε όλους τους τομείς όπου έχει η δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να αναφέρουν όχι μόνο τις παράνομες δραστηριότητες αλλά οποιαδήποτε παρατυπία. Η σημασία της δράσης τους ε, είναι μεγάλη. Ε, Πρέπει να τους προστατεύσουμε διότι διασφαλίζουν την προστασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στάνταρ αλλά και η ελάχιστη αυτή προστασία για τους καταγγέλτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε μια συνεπή και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Το κόστος ε, δεν θα εμποδιστε τα κράτη-μέλη από το να προχωρήσουν σε εθνική νομοθεσία. Να πούμε επίσης πόσο σημαντικά είναι τα κανάλια και οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Έχω ακούσει τις απόψεις των σκιωδών και πήρα και τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες για αυτό το θέμα. Είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι θα Υπάρχει συνένεση για τα κανάλια αναφοράς. Ε, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να δημοσιεύονται οι πληροφορίες στο κοινό από τους καταγγέλτες, γιατί καμιά φορά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν ε, σκεφτούμε το παράδειγμα του Ντοντούρα, ο οποίο ε, είναι σημαντικό παράδειγμα εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούσε εσωτερικά να αναφέρει το θέμα, γιατί ο ε, εργοδότης του βοηθούσε τους πελάτες ε, να, να φοροδιαφεύγουν. Στο τέλος λοιπόν αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια. Ε, κάτι που ήταν πολύ κακό για την προσωπική του προοπτική. Οι περισσότεροι καταγγέλτες αυτό κάνουν συνήθως διότι φαίνεται ότι είναι η μόνη επιλογή και αυτό πρέπει να το δούμε ως νομοθέτης. Επίσης πρέπει να να δούμε τι θα γίνει με την αρχή αντιστροφή του βάρους της απόδειξης ε, που ζητήθηκε στεναρά. Αυτοί που ε, καταγγέλουν δεν θα πρέπει να ζητείτε να αποδείξουν τα στοιχεία που ε, παρουσιάζουν, ε, διότι δεν υπάρχει δόλος. Επίσης, ε, θα ήθελα να μιλήσω για ένα εξάρτητο Ευρωπαϊκό Σώμα Προστασίας των Καταγγελτών. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, χρειάζεται τέτοιο σώμα για να έχουμε μια συνεπή προστασία των καταγγελτών που φέρνουν στο φως ε, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τους κανονισμούς των κρατών. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα ταμείο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προστατεύει με ανεξάρτητες νομικές συμβουλές και αποζημιώσεις ε, τους καταγγέλτες σε περίπτωση ζημιών λόγω της δημοσίευσης των πληροφοριών. Τέλος, ε, έχουμε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη από τα άλλα θεσμικά όργανα, ειδικά την Κομισιόν, που είναι εμβληματική παρουσία της ε, σε αυτό το θέμα για την προστασία των καταγγελτών. Ζητώ λοιπόν ε, τώρα να ακούσω και τη γνώμη των άλλων σχεδόν και να εργαστούμε καλύτερα στο τέλος ε, της ημέρας. Δίνω τώρα το λόγο στους σκιώδεις. Ο Φούλιο Ματρουσέλο δεν είναι εδώ, αλλά θέλει να πει ευχαριστώ στον Πρόεδρο και λυπάται που δεν μπορεί να παρουσιάσει προσωπικά τις ε, παρουσιάσεις, τις απόψεις του και με ευχαριστεί που τον ε, υποκαθιστώ και λέει ε, πρώτον ευχαριστεί την εισηγήτρια την κυρία Σκοτ Κέιτο για την επιτελεστή συνεργασία υπήρξαν βελτιώσεις μετά τη συνάντηση των σκιωδών αλλά υπάρχουν μερικά πολύ σημαντικά σημεία που ακόμη πρέπει να αντιμετωπιστούν ποια είναι τα κύρια θα πρέπει να αναφέρουμε στη συμβαστική Β της... Ε, όχι, είμαστε κατά της αναφοράς της ε, οικονομικές κρίσεις στην ε, συμβαστική Β και επίσης προτιμούμε τις τομεακές προσεγγίσεις από την οριζόντια. Επίσης το κείμενο αναφέρεται στην Επιτροπή Τάξε. Αυτό αφορά το συμβασμό G και δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Επίσης, υπάρχουν μερικές ε, πολύ γενικόλογες διατυπώσεις στην AIDS, μαζί και με την, ε, τον όρο το βάρος της απόδειξης. Η λέξη βάρος είναι υπερβολικά γενικόλογη. Για την συμβαστική M που προτείνει να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ανεξάρτητη Αρχή για να λαμβάνει πληροφόρηση από τους καταγγελτές, δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί αυτοί οι φορείς έχουν ε, πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες και δημιουργούν ε, ένα διχασμό μεταξύ ενωσιακής και εθνικής αρμοδιότητας. Δεν ε, με βρίσκουν σύμφωνους αυτές οι προτάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε επόμενες συναντήσεις για να το συζητήσουμε. Αυτά ήθελα να μας πει ο Φούλβιο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Όλι Λούντβιξον, ο οποίος είναι ο σκιώδης των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι θαυμάσια η έκθεση την οποία ε, εκπώνησε η Μόλι Σκοτ Κέιτο για αυτό το σημαντικό θέμα. Τώρα για τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Βασικό είναι να υπάρχει επαρκής προστασία των καταγγελτών πολλοί πραγματικά δεν καταγγέλουν τα κακό σκημένα γιατί φοβούνται ε, τις κυρώσεις που θα υποστούν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πολύ ανησυχητικό ότι διάφοροι πολίτες και δημοσιογράφοι τελικά σέρνονται στα δικαστήρια αντί να απολαμβάνουν επαρκούς νομικής προστασίας όταν δημοσιοποιούν πληροφορίες προς το κοινό συμφέρον. Είτε πρόκειται για νομιμοποίηση προϊόντων, προϊόντος εγκλήματος, είτε πρόκειται για φοροδιαφυγή. Αυτά είναι βασικά θέματα. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους καταγγέλτες. Και οπωσδήποτε θα συνέβαλε στην ε, περαιτέρω αποτελεσματικότητα και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα βελτιώνει και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Ένωση. Πρέπει λοιπόν να προστατευτούν και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός του. Τι σημαίνει καταγγέλτης. Η νομοθεσία αυτή θα έπρεπε να περιέχει και συγκεκριμένα μέσα, εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως για παράδειγμα οικονομικές κυρώσεις κατά των εταιριών και η υποχρέωση για τους κατακέλτες να διατηρούν ή να μπορούν να επανέλθουν στην εργασία τους. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν σωστή προστασία και θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή που να την διασφαλίζει. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και οι σωστές ε, δίωδη, η σωστή διάβλη για να γίνονται οι καταγγελίες και να δίδεται και σωστή ε, νομική πλαισίωση στους καταγγελτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση ούτως ώστε να έχουμε μια προστασία επαρκής ευρωπαϊκό επίπεδο των καταγγελτών και οριζόντια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλα, Λέω Πρόεδρος. ECR. Πύρκο Ρουόνεν Λένα είναι ο Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία. Η προστασία των κατακελτών μπορεί να φαίνεται ως ένα δευτερεύον θέμα στην πολιτική ίσονο σημασίας για την εργασία της ΕΚΟΝ, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι αν δεν είχαν υπάρξει οι καταγγέλτες και η τάξη και η πάνα δεν θα είχαν δημιουργηθεί. Δεν θα είχαν δημιουργηθεί. Και επίσης ε, και διάφορες άλλες ε, υποθέσεις δεν θα είχαν ε, δει το φως της δημοσιότητας. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους κατακέλτες γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Να υπάρχουν σαφείς ορισμοί και να υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία που να εγγυάται επαρκή προστασία. Θα μπορούσαν να προβλέπονται και οικονομικές παροχές, δηλαδή αποζημιώσεις ε, για παράδειγμα για δικαστικά έξοδα. Όπως θυμόμαστε και από την υπόθεση LuxLeaks, η προστασία των καταγγελτών στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Πρέπει λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα οι καταγγέλτες να καταγγείλουν τα κακό σκήμενα χωρίς να φοβούνται κυρώσεις. Υπάρχουν νομικά θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και το πώς εντάσσεται ε, στους εθνικούς ε, ποινικού κώδικες. Πρέπει λοιπόν αν υπάρχει πολιτική βούληση ή μάλλον καλύτερα αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να λυθούν τα ζητήματα αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη σοβαρές ανεπάρκειες. Δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα για να εγγυώνται την προστασία των κατακελτών. Γιατί ο τρόπος που παρουσιάζονται ορισμένα θέματα είναι ηθικά αφισβητήσιμος αλλά ορισμένε φορέ δεν είναι καθαρά παράνομα αυτά τα οποία καταγγέλνουν οι καταγγελτε. Στον... Στα κείμενα του ΟΣΑ υπάρχουν κάποιοι ορισμοί, αλλά είναι, δεν είναι επαρκώ ε, ε, ευρύ και άρα δεν έχουν ε, την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε φορά που συζητάμε την ε, φοροδιαφυγή ή την ανάγκη να υπάρχουν δημόσια μητρώα για τους ε, πραγματικούς δικαιούχους των εταιρεών, να συζητάμε και τα θέματα των καταγγελτών ακριβώς εκείνων που δεν σέβονται αυτά τα μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν σωστοί διάβλοι για να μπορούν να ε, καταγγέλουν τα κακοσκήμενα οι καταγγέλτες και οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να τους παρέχουν προστασία. Εξάλλου και οι ίδιες θα προστατεύονταν από την δραστηριότητά τους τελευταία ανάλυση και θα λειτουργούσαν καλύτερα. Εάν καταφέρουμε να ε, διευρύνουμε τον όρο, δεν πρέπει να πούμε απλώς ε, ε κείμενα σε, στο δημόσιο τομέα. Οι τροπολογίες πηγαίνουν προς την κατεύθυνση και ελπίζω να επιτευχθεί σύντομα πρόοδος. Ωστόσο πρέπει να βασίσουμε την εργασία αυτή σε, νομικό, σε σωστό νομικό έλεγχο για να μην έχουμε προβλήματα αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πύρκο, για τους φιλελευθέρους. Δεν βλέπω όμως κανένα φιλελεύθερο εδώ. Καλώς. Κούε. Ο κύριος Παπαδημούλης. Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Μόλι Σκότ για τη δουλειά που έχει κάνει και το χρόνο και την ενέργεια που έχει αφιερώσει ε, στο συγκεκριμένο φάκελο. Ε, το σχέδιο που έχει παρουσιάσει από την αρχή είναι θετικό, επιδιώκει να συγκροτήσει μια γνωμοδότηση με ένα σχέδιο ισορροπημένο και σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που έχει θέσει η πραγματικότητα γύρω από το θέμα της προστασίας των καταγγελτών, των whistleblowers. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η προστασία των whistleblowers είναι ανεπαρκής και χρειαζόμαστε μία πανευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας των whistleblowers, γιατί αυτό υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε εκτεταμένα προβλήματα, παραβίασης της νομιμότητας, διαφθοράς φοροδιαφυγής, είναι να θωρακίσουμε το πλαίσιο όσων επιδιώκουν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, αποκαλύπτοντας εμπιστευτικές πληροφορίες ιδιωτικών επιχειρήσεων ή και δημόσιων οργανισμών. Η έκταση του προβλήματος είναι μεγάλη, το μέγεθος της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς είναι μεγάλο και δυστυχώς έχουμε μέχρι τώρα φαινόμενα όπου αντί να τιμωρηθούν οι παραβάτες της νομιμότητας που κλέβουν το Δημόσιο Ταμείο και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρούνται όσοι αποκαλύπτουν την παρανομία και την παράβαση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα οθήσει και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη δική τους νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία των καταγγελτών. Και αυτό νομίζω ότι υπηρετεί όχι την προστασία μόνο των whistleblowers, αλλά τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου. Ένα τέτοιο αναβαθμισμένο πλαίσιο θα επέτρεπε σε περισσότερους να τολμούν να αποκαλύπτουν πληροφορίες που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και που σήμερα φοβούνται να το κάνουν γιατί κινδυνεύουν να βρεθούν οι ίδιοι κατηγορούμενοι και να υποστούν ποινές, διώξεις, φυλακίσεις, εκβιασμούς. Νομίζω ότι οφείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι πάντες και οι μεγάλες εταιρείε οφείλουν να σέβονται τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου, τις κοινωνίες, τους φορολογούμενους πολίτες που υπερφορολογούνται, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι, για να φορολογούνται αυτές μέσω παράνομων πρακτικών ελάχιστα. Οι συμβιβαστικέ τροπολογίες που έχει καταθέσει η συνάδελφο μόλις Σκότ, κατά τη γνώμη μου, κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Σε κάποια του σημεία εμείς θα θέλαμε πιο τολμηρές και πιο ε, σαφείς αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια ευελιξία εκ μέρου του εισηγητή για να εξασφαλιστεί η ε, ευρύτερη δυνατή συνένεση και ένα κλίμα σύνθεσης ε, που να εξασφαλίσει ευρεία στήριξη. Το ίδιο θα ήθελα και από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σε ένα μόνο σημείο επιτρέψτε μου να αναφερθώ. Ε, η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των καταγγελτών πρέπει να συνδεθεί και με κοινέ πολιτικές που αναπτύσσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η παγκόσμια κοινότητα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να, να συμπεριλάβουμε, να λάβουμε υπόψη μας σε αυτή τη γνωμοδότηση, έστω και στα recitals, το άρθρο 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ εναντίον της διαφθοράς. Είναι σημαντικό η προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή μας και όλο το Ευρωκοινοβούλιο να συνδεθεί με τις μέχρι τώρα προσπάθειες και άλλων θεσμών και διεθνών οργανισμών. Με αυτό το πλαίσιο θα στηρίξουμε την εισήγηση της ε, συναδέλφου Μόλι Σκότ και πιστεύω ότι και το απόγευμα θα επιτύχουμε μια ευρεία συνένεση. Σας ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον εκπρόσωπο της UFTD. Ε, δεν έχω κανένα στον κατάλογο μου ε, που ζητά τον λόγο. Ωραία. Τότε σταματάει ο πρόεδρος. Ξέρεις για ποιο θέμα μιλάμε. Είναι ναι, Πρόεδρε, πιστεύω πως ε, συζητάμε τους ε, καταγγέλτες. Θέλω να θέσω μια ερώτηση σύντομα στην ε, Μόλη για να δω αν αντιμετωπίζει το θέμα της, των πόρων ώστε να υπάρχει ένα κονδύλι, ένα ταμείο για τους καταγγέλτες γιατί διαφορετικά είναι, αρκε... είναι δύσκολο συχνά να έχουν πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη με την κατάλληλη νομική ε, στήριξη. Ήθελα να ξέρω λοιπόν εάν υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι για τους καταγγέλτες. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Για να απαντήσω στην ερώτηση της Νίνα, υπήρξε μια τροπολογία που ζητούσε την δημιουργία ενός ταμείου για την προστασία των καταγγελτών. Εγώ συμφωνώ πως είναι πολύ σημαντικό, είναι τεράστιο έργο, ενώ οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται συχνά με χαμηλό μισθό. Μπορεί δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλουν ε, σημαντικά δικαστικά έξοδα να τους αποτρέπει από το να γίνουν καταγγέλτες, γι' αυτό και σκεφτόμαστε το να συμπεριλάβουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου στην πρόταση που υποβάλλουμε. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, είπατε ότι η οδηγία ε, για την, το ξέβλημα χρήματος είναι προτεραιότητα για μας και σε αυτή την περίπτωση τον έχουμε πληροφορίες πληροφορίες για το πότε γίνεται ξέπλυμα χρήματο ή πότε υπάρχει φοροαποφυγή είναι πολύ σημαντικό για εμά του νομοθέτες για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τι ε, κακέ αυτέ πρακτικέ Είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσονται αυτέ οι πληροφορίε, σημαντικό στοιχείο στα δημοκρατικά συστήματα και γι' αυτό και προσπαθούμε να στήσουμε την πιο καλή προστασία για αυτού του ανθρώπου. και είναι η ευκαιρία για να στηρίξουμε αυτή μα τη θέση προ την Κομισιόν για το είδο τη νομοθεσία που θα πρέπει να έχουμε σε ολόκληρη την Ένωση για να προστατεύουμε του καταγγελτέ. Έχουμε έναν καλό βαθμό δέσμευση όσον αφορά τη σημασία αυτού του φακέλου και καλό βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη για να το καταφέρουμε. Οπότε θα έχουμε μάλλον επιτυχή συνεδρίση και προσβλέπω να σας ξαναδώ και το απόγευμα ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσουμε αυτό το, αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη διαπραγματευτική ομάδα που θα συνεδριάσει απόψε ε, για τον επόμενο γύρο για τη βελτίωση των συμβιβαστικών. Προβλέπεται η ψηφοφορία στις 4 Σεπτεμβρίου την επόμενη εβδομάδα και η επί της ουσίας, ε, αρμόδια επιτροπή, η νομική, θα ψηφίσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την εργασία μας λοιπόν, εάν θέλουμε να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μας από την ε, Νομική Επιτροπή. Φτάνουμε στο σημείο 6 που είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018 όλα τα τμήματα εισηγητής είμαι εγώ. Οπότε παίρνω το λόγο και αν συμφωνείτε θα μιλήσω στην γλώσσα μου, δηλαδή στα γερμανικά. Όταν είναι κανείς από τη Βαβαρία δύσκολα μιλάει καλά γερμανικά, αλλά θα το προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν 60 τροπολογίες ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης που έχω καταθέσει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των συναδέλφων και είναι καλό που υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Εχθές ε, το απόγευμα έγινε μια συνάντηση των σκιωδών και εκεί ε, ε, βρήκαμε 7 συμβαστικές τροπολογίες, τις δουλέψαμε εχθές και ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση για αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες στην ουσία συνοψίζουν ένα μεγάλο κομμάτι των 60 αρχικών τροπολογιών. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τις προτάσεις και την επικοδομητική συνεργασία, ε, γιατί πάντοτε όλα πρέπει να πάνε μεταξύ τέλη Αυγούστου, τελών Αυγούστου και αρχών Σεπτεμβρίου πολύ γρήγορα. Ε, να πω ότι για μένα ένα θέμα που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ε, ήταν ε, η εντολή των Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας αλλά και οι επιπτώσεις του Brexit στην εργασία μας ειδικά, στις εργασίες τους, ειδικά σε μία από αυτές τις αρχές. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε τον προϋπολογισμό για τις τρεις αυτές αρχές. Ε, ε, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένας σωστός προϋπολογισμός και να έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε αυτές τις τρεις αρχές και τον προϋπολογισμό τους, διότι παραδοσιακά ε, ήταν, ήταν πάντοτε σημαντικό ε, να γνωρίζουμε και τις ε, προτάσεις της Κομισιόν για αυτό το review. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει γενικά ομοφωνία ότι αποτελούν αυτές οι αρχές, αρχές συντονισμού και εποπτείας και θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα κονδύλια για να δρουν ούτως. Είναι σημαντικό λοιπόν να δίνουμε τα κονδύλια μας ε, στοχευμένα και οι νομοθέτες ε, πρέπει να το κάνουν αυτό με βάση τις αντίστοιχες εντολές. Θα πρέπει λοιπόν στην πράξη αυτό να μεταφραστεί και θα πρέπει ε, να δούμε ότι δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν τηρήθηκε. Το ΜΥΦΙ 2, για παράδειγμα, ήταν ε, κάτι ε, στο οποίο είχαμε προτάσεις παρά ε, τη θέληση, ας πούμε, του, την αρχική θέληση του νομοθέτη. Νομίζω λοιπόν ότι το η πολιτική εντολή εδώ, αυτή που είναι στην οδηγία, στην ουσία, ε, μειώνεται σημαντικά από τις προτάσεις της ΕΜΠΑ τις αρχές για την Τράπεζα. Λοιπόν, ε, θα πρέπει εμείς ε, είτε τελικά να αγνοούμε, φαίνεται ότι είτε τελικά αγνοείται η εντολή που δόθηκε από τον νομοθέτη, είτε χρησιμοποιείται λανθασμένα. Θα πρέπει λοιπόν να, παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν, έτσι ώστε να δούμε αν αυτά τα παραδείγματα είναι μεμονωμένα ή ε, αν θα πρέπει να στείλουμε ε, κάποια προειδοποίηση σε αυτές τις αρχές ώστε να ε, δρουν διαφορετικά. Τώρα για το Brexit, οι επιπτώσεις του για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης θα φέρουν πολύ φόρτο εργασία στις τρεις αρχές. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρχές αυτές μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση των, του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα μία από τις αρχές που έχει την έδρα της στο Λονδίνο θα πρέπει να μεταφερθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις, το κόστος για παράδειγμα. Ε, χωρίς ε, το Brexit δεν θα υπήρχε ε, κόστος και με το Brexit υπάρχει. Υπάρχει σχετική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να φέρει το κόστος για αυτή την μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών από το Λονδίνο. Η επόμενη, η υπόλοιπη 27 Βέβαια, αναρωτιόμαστε πού θα πάει αυτό, αυτή η αρχή. Αυτό ε, δεν θα το αποφασίσουμε όμως εμείς, αλλά θα το επικυρώσουμε. Καλό θα ήταν ε, να έχουμε κάποια στοιχεία, να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη αποτελεσματικότητα και να βελτιώσουμε το κόστος. Είναι τρεις μικρές αρχές, οι οποίες όμως θα πρέπει ε, να φέρουν το φόρτο της εργασίας ε, που είναι μεγάλος. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι σε κάποια σημεία θα πρέπει να ρίξουν περισσότερη δουλειά. Και αυτό φαίνεται και στις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Να δούμε αν θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε κάποιες από αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια και να δούμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Επίσης, ε, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο κόστος ενοικίου των ε, γραφείων των αρχών αυτών. Ε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η ΕΙΟΠΑ στη Φραγκφούρτη πληρώνει τη μισή τιμή τετραγωνικό από ό,τι πληρώνουμε στο Παρίσι. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία δυστυχώς, αλλά στην διαδικασία του προπολογισμού αυτά τα ελέγχουμε. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει και εκεί χώρος ε, για να εξοικονομήσουμε κονδύλια. Ίσως στο μέλλον λοιπόν ε, καλό θα ήταν και για την EBA και για την ΕΙΟΠΑ να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεκονομήσουμε κόστος ε, από το ενίκιο. Γιατί και στο Λονδίνο ήταν ψηλά τα ενίκια, όπως είναι και στο Παρίσι, όπου βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Αρχή. Ε, αλλά θέλω λίγο να τα συζητήσουμε αυτά. Νομίζω ότι με τις 7 τροπολογίες στην ουσία ε, καλύπτουμε όλες τις προτάσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ για την επικοδηματική συνεργασία και χαίρομαι για την ε, συζήτηση. Θα γυρίσω τώρα στα αγγλικά γιατί είμαι και πάλι πρόεδρος. Πρώτος είναι ο Όλι Λούντιξον ο σκιώδης από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέρμπερ για τη σύντομη και περιεκτική έκθεση. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το να χορηγηθούν πόροι στις αρχές ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Η συζήτηση για το μέλλον της ΟΝΕ είχε ζωηρέψει πριν το καλοκαίρι και πιστεύω πως αυτό ήταν πολύ καλό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν επαρκείς πόροι και για αυτό το σκοπό. Το Συμβούλιο, ωστόσο, έχει περικόψει αυτή τη γραμμή του προπολογισμού και εγώ ε, και οι εισηγητής θελήσαμε να αποκαταστήσουμε, να επαναφέρουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν, ώστε να υπάρχουν ε, επαρκείς πόροι για την επιβίωση της ε, ΟΝΕ. αυτό θα ήταν λογικό, πιστεύω, να συμπεριληφθεί και στην γνωμοδότησή μας την οποία αναφέρω στην τροπολογία μου. Στην γνωμοδότηση υπάρχει ένα κείμενο που λέει για την ε, σταθμισμένη, ε, ε, σταθμισμένους πόρους για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ευρύτερα κάτι, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην θέσουμε σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της αρχής, του οργανισμού αυτού, γιατί ε, μπορεί αυτή η φάση να αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι κατά δε του να βάλουμε την ε, EBA μαζί με τις άλλες, τους άλλους οργανισμούς γιατί αυτή η, αυτός ο οργανισμός προσπαθεί και δυσκολεύεται να βρει την σωστή ισορροπία ε, ανάμεσα στη συμφέροντα και την εφαρμογή της νομοθεσίας δευτέρου επίπεδου. Ο στόχος μας είναι να είναι πιο αποτελεσματική η αρχή αυτή και επίσης θα πρέπει να προστατεύονται οι καταναλωτές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι οποίοι συχνά ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την ενημέρωσή τους αν τη συγκρίνουμε με τους ε, τραπεζίτες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γι' αυτό και πρέπει να προστατευτούν. Επίσης θέλω να τονίσω τη σημασία της ολοκλήρωσης της εργασίας των εργασιών μάλλον της Κομισιόν για την ε, ε, Ένωση των ε, Κεφαλαγορών αλλά και για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα είναι αυτό πολύ σημαντικό για την αγορά αυτή και θα είναι επίση σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Μεγάλο κομμάτι δε των ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να αφιερωθεί στην καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή αλλά και του επιθετικού φορολογικού, φορολογικού σχεδιασμού. Και γι' αυτό και αναφέρομαι στην αποκατάσταση, στην επαναφορά της αρχικής πρότασης της Κομισιόν όσον αφορά τη βελτίωση του φορολογικού συστήματο και τη στήριξη των προπαρασκευαστικών μέτρων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί νομίζω και στην γνωμοδότηση. Να επαναλάβω δε ότι όπως και ο εισηγητή πιστεύω πως το επιπλέον κόστος που προκαλείται από τη μετακίνηση της EBA ε, της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής θα πρέπει να ε, επιβαρύνει αποκλειστικά την Βρετανία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία σας και για το ότι θελήσατε να λάβετε υπόψη τις ιδέες μου και να φτιάξουμε έτσι συμβαστικές ε, προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ όλε. Η Μπίργκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις συμβιβαστικές και για τις ε, περιστατωμένε συζητήσει. Εκ μέρου του κ. Λούντ θέλω να σα ενημερώσω ότι συζητηρίζουμε όλες τις συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό μόνο ήθελα να ακούσω. Από τους φιλελεύθερους έχουμε τον κύριο Τόρβαλτ, αλλά δεν ε, έχει έρθει. Οπότε έρχομαι στην Γκούε που έχουμε τον Μιγγέλ Βιέρας Βιέγα, συγγνώμη, που επίση λείπει και ο μοναδικό εκπρόσωπο τη ΓΚΟΕ ε, μας εγκαταλείπει, οπότε Σβέν, εσύ τώρα έχει το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για τη σχέδια έκθεση και για την κάλυψη των τροπολογιών από τον εισηγητή. Είμαστε ευχαριστημένοι για το πώς προχώρησαν τα πράγματα. Απλά θέλω να εκφράσω μια επιφύλαξη και αυτή αφορά την διατύπωση της συμβιβαστική που μας που, μας, που μιλά για τους εποπτικούς οργανισμούς, γιατί ε, έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά πάντοτε αυτοί ενεργούν στο πλαίσιο που εμείς έχουμε θεσπίσει ως συνομοθέτες, στο πλαίσιο της εντολής τους προστασία καταναλωτή και έχουν καλύψει διάφορα κενά και επίσης πρέπει να εξασφαλίσουν την συνεπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό εντάσσεται στον κανονισμό των τριών εποπτικών αρχών. Τώρα μπορεί να υπάρχουν πολιτικές αποκλήσεις κατά που κανείς στηρίζει αυτά τα μέτρα ή όχι, είτε μήπως ήταν υπερβολικά. Πάντως ήταν εντός των εντολής. Αυτή είναι η οχι η μηπως ηταν υπερβολικα παντως ηταν εντος επιφύλαξη και θέλω επίσης να πω στον Όλε ότι δεν μ' αρέσει να διαφωνώ μαζί σου, αλλά όσον αφορά την EBA και την ΑΙΟΠΑ, το Κοινοβούλιο ανέκαθεν, όπως και η συγητής, στήριξε η το ότι αυτές οι υποπτικέ αρχές θα πρέπει να είναι μαζί, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη δεν γίνεται συστηματική διαφορά ανάμεσα στις ασφαλιστικέ και στις τραπεζικές εταιρείε. Έχουμε τεράστιε ομίλου. άρα η ΕΚΤ δεν έχει ευθύνη. Ακόμα και αν εποπτεύει μια τράπεζα ή κάποιον φορέα που, κάνει ασφαλίσεις και τραπεζικές ε, ε, δραστηριότητες. Γι' αυτό και η ΕΜΠΑ και η ΕΙΟΠΑ ποτέ δεν θελήσαμε να είναι σε δύο διαφορετικές πόλεις. Το Κοινοβούλιο ήθελε να είναι όλοι μαζί σε ένα μέρος. Γι' αυτό και ο εισηγητής πρότεινε να προχωρήσουμε σε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον εκεί που υπάρχει μεγάλη επικάλυψη ανάμεσα στις ασφαλιστικές και στις τραπεζικές δραστηριότητε. Ανδιάφορο το πού θα είναι αυτή, ποια θα είναι αυτή η πόλη. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, θα γίνουν πολλές συζητήσεις με το Συμβούλιο όσον αφορά αυτό το στοιχείο. Το θέμα αφορά το, το μέρος, την τοποθεσία, που για μας είναι ε, δευτερογενές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε κάτι το διά. Είναι ένα γκίλ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καλό είναι που μπορούμε να συζητήσουμε προϋπολογισμούς, γιατί έχουμε συζητήσει συχνά προϋπολογισμούς. Για αυτούς τους υποπτικούς οργανισμούς, το βασικό είναι να υπάρξει πιο αποτελεσματική λειτουργία και επίσης να βρούμε και άλλους πόρους για αυτές. Καλά λοιπόν τα λένε συμβασμοί DKE. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όμως για την πρότασή σας για την ε, τραπεζική αρχή, το EBA, ότι θα πρέπει να πληρώσει το Λονδίνο το κόστος. Με ακούτε πρόεδρε. Α. Είναι πρόωρο πιστεύω να κάνουμε αυτή τη διατύπωση γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις. Και ήδη υπάρχει μια συζήτηση για το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και σίγουρα θα συμπεριληφθούν και τα θέματα αυτής της ε, μεταφοράς της EBA στις διαπραγματεύσεις. Άρα είναι πρόωρο. Είναι πραγματικά πρόωρο. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποχωρήσει από την ενιαία αγορά τι ακριβώς θα διαπραγματευτούμε τότε. Νομίζω ότι είναι πρόωρο για το 2018 το θέμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Έχω λοιπόν πολύ ισχυρές επιφυλάξεις για τη συμβαστική ΕΦ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Να ξαδώσω το λόγο στον συγκητή, ο οποίος θα ξαναμιλήσει γερμανικά. Με συγχωρείτε, ε, είμαι εδώ με δύο καπέλα. Καταρχάς λοιπόν ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ξέρω ότι κάθε ομάδα κάνει ό,τι μπορεί. Και το βασικό είναι να κάνουν όλοι υποχωρήσεις για να επιτευχθεί σωστό συμβασμός. Και το επιχειρήσαμε χθε και νομίζω ότι επιτύχαμε και χάρηκα ιδιαίτερα που οι σοσιαλιστές για το θέμα της συγχώνευσης ε, των οργανισμών υπήρξε καλή θέληση για να συμπεριληφθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει υποστήριξη τουλάχιστον από τους σοσιαλιστές για την πρότασή μου και ανάγκη περαιτέρω συζήτησης. Και για άλλα θέματα υπάρχει ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ τον Όλε που επίσης ε, ανέφερε τα θέματα που υπάρχει συμφωνία σε, με λεπτομέρειες. Ε, αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες γραμμές του υπερπολογισμού. Για το θέμα τώρα του κόστους να τολμήσω να πω ότι ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Απρίλιο του 19 παραμείνει στην ε, ενιαία αγορά, κάτι που δεν νομίζω ότι είναι η εντολή που έχει αναλάβει από μόνη της η Βρετανική κυβέρνηση, παρόλα αυτά θα θεωρούσω ότι δεν είναι δυνατόν να παραμείνει εκεί ευρωπαϊκός φορέας. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες νομικές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα για το θέμα του εάν και κατά πόσο θα είναι ακόμη ε, εντός δικαιοδοσίας το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί επιχειρεί, όπως ξέρετε, να ε, αποχωρήσει και από την ε, δικαιοδοσία του δικαστηρίου και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η τραπεζική αρχή θα είναι εκτός δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ε, υπόθηκε εκτός μικροφώνου ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα μεταβατικό καθεστώς. Ζήτησα όμως να μάθω μέχρι πότε είναι η μίσθωση της ε, ΕΜΠΑ και δεν, είναι τόσο, ε, δεν πάει τόσο μακριά όσο η μίσθωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς μεταβατικές ρυθμίσεις θα υπάρξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη φύση των πραγμάτων αλλά είναι ένα θέμα όπου μόνο μέσω της ψηφοφορίας θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συνένεση ή όχι. Νομίζω ότι μέσω λοιπόν δημοκρατικής διαδικασίας, δηλαδή μέσω ψηφοφορίας, θα καταλήξουμε από αυτού. Από ό,τι κατάλαβα από ό,τι είπαν οι άλλες πολιτικές ομάδες, υπάρχει ευρεία συνένεση γι' αυτό. Η ψηφοφορία θα είναι σήμερα το απόγευμα. Παρακαλώ να είστε όλοι παρόντες με τις κάρτες ψηφοφορίας για να μην έχουμε προβλήματα. Η διαδικασία προβλέπει ότι αυτή τη βδομάδα θα πρέπει να εγκρίνουν όλες οι επιτροπές τις γνωμοδοτήσεις τους για τον προπολογισμό, ούτως ώστε μετά η Επιτροπή Προπολογισμών ε, με τα λόγου γνώσεως να προωθήσει γενικά το θέμα του προπολογισμού, να το αποφασίσει εντός του Σεπτεμβρίου και μετά η ψηφοφορία στην Ολομέλη να γίνει τον Οκτώβριο όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Τώρα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με βάση λοιπόν την ημερήσια διάταξη, περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι το 8. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το φόρο προστιθέμενης αξίες για ε, παραγωγές υπηρεσιών και πωλήσει αγαθών εξ αποστάσεως. Έχουν οι σοσιαλιστές κάποια πληροφόρηση για το πότε θα έρθει ο εισηγητής. Θέλετε να έχουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11. Ωραία, διαλυματάκι μέχρι τις 11. Φαίνεται ότι τα τελειώσαμε όλα πριν ε, από την ώρα τους, αλλά ξεκινήσαμε ένα λεπτό μετά τις 10. Άρα, διάλειμμα μέχρι τις 11.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

Okay.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 Thank

Σύμφωνα με το ρολόι, η ώρα είναι τώρα 11. Συνεχίζουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξή μας. Είμαστε στο σημείο 8 και 9. Μαζί θα τα εξετάσουμε. Ξεκινούμε λοιπόν με τον εισηγητή για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσει αγαθών εξ αποστάσεως. Είναι ο Καταλίνος Σόριν Ιβαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει. Η πρόταση της Επιτροπής ε, είναι για ένα πακέτο είναι η απάντηση της Κομισιόν για το σύστημα ΦΠΑ. Είναι μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του συστήματος ΦΠΑ. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα εδώ. Ε, η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται στο ΜΟΣ, ε, τη μικρή μονοαπευθυντική θηρίδα, η οποία εισήχθη για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια επιτυχία, διότι μειώνεται ο διοικητικός αλλά και επειδή αυξήθηκαν τα έσοδα του, των, του κράτους. Θέλουμε λοιπόν να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής ε, του ΜΟΣ της μικρής μονοαπευθυντικής θηρίδας, ε, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη χρήση. Κυρίως ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να απλουστεύσουν τις διαδικασίες τους. Χαιρετίζω λοιπόν την τροποποίηση του άρθρου 28 που ζητά από τις ε, επικραμμικές ε, πλατφόρμες ε, να αναλαμβάνουν την ίσπραξη του ΦΠΑ. Όμως πολλές φορές επειδή αυτές οι πλατφόρμες είναι διάμεση κατά την προμήθεια αγαθών από τρίτες χώρες, βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες τελικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις ε, εταιρείε από τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές υπηρεσίες χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ. Για να βιαλτιώσουμε λοιπόν την ίσπραξη του ΦΠΑ και να απλουστεύσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε προχωρήσει σε, αυτή... σε αυτό το βήμα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες ε, οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην ουσία υποστηρίζουν αυτά που ήδη ανέφερα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τους συναδέλφους τις απόψεις τους. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έβρασης συνένεσης, τουλάχιστον στη συνάντηση των σκιωθών ε, που θα έχουμε στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή τη συνένεση. Υπάρχει ε, κάποιο όριο, ε, το λεγόμενο όριο των 10.000 ευρώ, που υπάρχουν κάποιες διαφορές γι' αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι θα υπάρξει συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Πάμε στο σημείο 9, που είναι η διοικητική συνεργασία για καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο Λούντεκ Μάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Μάρκους. Είναι μια ε, συνδιαλλαγή που έχει να κάνει και με την έκθεση του Ιβάν έχει να κάνει με την υποδομή και τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να επεκταθεί το μόσες της ε, πωλήσει εξαποστάσεων, αγαθών εξαποστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από τεχνική άποψη λοιπόν, εδώ έχουμε πιο απλή υπόθεση, έχουμε 22 τροπολογίες, ε, οι τέσσερις από αυτές όμως δεν είναι αποδεκτές. Επίσης, φαίνεται ε, ότι υπάρχουν τροπολογίες που λένε ότι θα πρέπει η εφαρμογή να πάει από το 2021 το 2019, να γίνει πιο γρήγορα δηλαδή. Ήρθαμε όμως σε επαφή με την Κομισιόν η οποία μας είπε ότι τελικά η ημερομηνία που προτείνανε υποδεικνύεται από την ε, ιδιαίτερα περίπλοκη τεχνική φύση του συστήματος. Δεν θα είναι εύκολο λοιπόν να γίνει νωρίτερα, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα ε, για τις εταιρείε. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να μείνουμε με την αρχική πρόταση. Όπως και να έχει, σύντομα θα ψηφιστεί η έκθεση και θα ε, αξιολογηθούν αυτές οι 22 τροπολογίες. Δεν θα είναι περίπλοκη ψηφοφορία. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε τον Λούντεκ. Πάμε στους Κιώδης. Ξεκινάμε με τον Βέρνερ Λάγκεν από το ΕΛΚ. Κάτι σύντομο για την ε, μοναπευθυντική θηρίδα για τις διαμεθοριακές ε, συναλλαγές. Υπάρχουν 39 ε, τροπολογίες, είναι κυρίως τεχνικές, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το μόνο επίμαχο σημείο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι το ανώτατο, το, η τιμή κατοφλίου για να, για να υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή είναι 100.000. Η Κομισιόν προτείνει να κατέβει 10.000 για να μην υπάρχει στρέβλωση τη αγορά. Αυτό είναι το νόημα του προγράμματο για το ΦΠΑ γενικά. Θεωρώ ότι γένεια η μείωση αυτού του κατοφλίου και σωστά την αιτιολογεί η Κομισιόν. Οπότε θεωρώ ότι οι τροπολογίε Σκοτ Κάτου των φιλελευθέρων που δεν θέλουν να αλλάξει το όριο αυτό ή τη κυρία Νίνιουζεν και του ECA, του Μπέντ Λούκε, που λέει να πάει στα 35.000 θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι τροπολογίες δεν είναι καλύτερες ε, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Νομίζω ότι με μόνο μία συνεδρίαση των σχεδόν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές που προετοίμασαν με τόσο εύληπτο τρόπο τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος για τους σοσιαλιστές. ο κύριος Φρουντσούλητσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης για την εργασία τους για αυτό το σημαντικό θέμα. Γιατί είναι σημαντικό τμήμα του πακέτου νομοθεσίας για τον ΦΠΑ που είναι σημαντικός πόρος για τα κράτη-μέλη και βοηθάει και την ανάπτυξη αν χρησιμοποιηθεί σωστά βέβαια. Η πρόταση αυτή μας βρίσκει σύμφωνους. Σύμφωνη, μάλλον σέβεται τις αρχές της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Είμαστε λοιπόν πλήρως υπέρ της ε, έγκρισης της. Θέλουμε να διευρυνθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την μίνι απευθυντική θηρίδα θα έχει θετικές ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις και συμφωνώ και με την πρόταση του συγητή να έχει πρόσβαση η Επιτροπή μόνο στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για λόγους στατιστικής. Να μην υπάρξει δηλαδή υπερβολική γραφειοκρατία προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εξαγάγουν τα σωστά στοιχεία. Οπότε, η επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και κομισιών θα πρέπει να είναι επαρκής και αποτελεσματική, ούτω ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ε, της, ε, του κανονισμού εγκαίρως. Επίσης να δούμε σε τι βαθμό θα μπορούσαν να εφαρμοστούν είτε η μία ή και οι δύο, μάλλον είτε ο ένας είτε και οι δύο κανονισμοί πριν το 2021 ένα πρώτο βήμα για να λάβουμε υπόψη την ταχεία εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει οι κανόνες για το ΦΠΑ να περιορίζουν την επέκταση της ε, οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, οι σκιώδεις ε, θα αναφερθούν και στις δύο εκθέσεις, ECR ε, πρώτα και τους δύο. Ευχαριστώ. Καλό είναι να τις συζητήσουμε μαζί και τις δύο προτάσεις. Σε προηγούμενες συζητήσεις σας έχω παρουσιάσει την άποψή μου και για τις δύο προτάσεις αυτές. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που έχω ήδη πει. Νομίζω ότι θα πάνε καλά αυτές οι προτάσεις. Ούτε οι τροπολογίες θέτουν ανυπέρβλητα προβλήματα. Συμφωνώ με την ε, εκτίμηση του κύριου Μπενλάγκε ότι με μια συνεδρίαση των ε, σκιωδών θα ε, επιλύσουμε τα θέματα για το κατόφλιο για αυτές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί τώρα 35, 10, καλά δεν είναι ότι είναι απόλυτα ε, καθορισμένη η απόψή μου. Το θέμα είναι να μην υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Το βασικό είναι να μπορούν να υποφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Νομίζω ότι στη συνεδρίαση των, συντονιστών, σκιωδών θα το επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Ε, Λίμπε Βέρινγκ. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εκ μέρους ε, της Κόρο. Αυτή η νομοθεσία θα ενισχύσει την ενιαία αγορά απλουστεύοντας τους κανόνες και διευκολύνοντας ε, την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, θα σταματήσουν οι εξαιρέσεις για τους ε, μη Ευρωπαίους ε, και θα επεκταθεί η μικρή μονοαπευθυντική θηρίδα. Θεωρώ λοιπόν ότι με την Κομισιόν συμφωνούμε για αυτή την πρόταση όμως θα ήθελα να τονίσω ότι οι επιπτώσεις τουλάχιστον για τον τομέα των ταχυδρομικών και υπηρεσιών και υπηρεσιών courier χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι πωλήσει εξ αποστάσεων, εξ ειδικά ε, από τρίτες χώρες ε, έχουν μεγάλη επιβάρυνση για τους υποκείμενους σε φόρο. Ε, ειδικά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι μικρές αποστολές έως και 150.000 ευρώ θα οδηγήσει σε λιγότερο διοικητικό κόστος. Γι' αυτό προτείνω τα όριο, το ελάχιστο όριο που αναφέρθηκε προηγουμένως από τα 10.000 ευρώ δηλαδή να καθοριστεί στα 35.000 ευρώ διότι έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια με τις τρέχουσες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Αδειμονώ λοιπόν για μια συμβαστική λύση και ελπίζω να εγκριθεί η νομοθεσία αυτή χωρίς ε, καθυστέρηση. Για το σημείο 9 η Κόρα λέει ότι ε, αυτό το σχέδιο που κατατέθηκε πριν το καλοκαίρι στην ουσία με κάνει ένα για την εφαρμογή του άμεσα. Θα έχει μια θετική επίπτωση στα εξόδα, τα κρατικά έσοδα και θα βελτιώσει ε, πάνω από 2 δις αυτά τα έσοδα. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Οι τροπολογίε που έχει ήδη προτείνει ο εισηγητής ε, είναι πράγματα που θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω με την πάταξη της απάτης και με ένα εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει να εντοπίζουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν απάτες μέσω διαδικτύου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του εργαλείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό ε, να χρησιμοποιηθεί αυτό το στοχευμένο εργαλείο από τις νόμιμες επιχειρήσεις για να μειωθούν και τα μέτρα κατά της απάτης. Ε, καλό θα είναι να πειραματιστούμε λοιπόν με αυτό και αδίμονο να δω ε, ποιες είναι οι συμβαστικές τροπολογίες και να δω να υιοθετείται η έκθεση. Πάμε τώρα στις σκιώδες από την ΚΟΕ, Παλώμα Λόπες, Μίγκουελ Βιέγκας. Δεν μπορώ να τους δω στην αίθουσα, οπότε πάμε στους πράσινους. Ε, Σκοτ Κέιτο δεν είναι εδώ, Μπάρμπαρα Κάπελ από το ΙΕΝΕΦ, e ούτε αυτή είναι εδώ. Δεν βλέπω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, όχι. Άρα επαναρχόμαστε στους εισηγητές. Ο κύριος Ιβάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ιδέα είναι απλή. Δεν έχουμε τα ζητήματα να συζητήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ειλικρινά ότι στην πρώτη συνάντηση σκιωδών στο Στρασβούργο θα επιλύσουμε όλα τα προβλήματα. Και ότι η έκθεση θα τύχει πλήρους συνένεσης. Άρα, δεν υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που χρήζουν συζήτησης και είμαι πεπισμένος ότι σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Λούντεκ, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ήσασταν πολύ γρήγοροι. Έχω το εξής πρόβλημα. Ο επόμενος εισηγητής, ο Ροβέρτο, δεν είναι εδώ, άρα και πάλι μέχρι τις 11.30 θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα.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

So, hello everybody. The Χαίρετε. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι ο εισηγητής μας ε, είναι ακόμη καθοδόν, αλλά δεν είναι ακόμη στο κτίριο. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με το 7, η έγκριση ορισμένων νομικών πράξεων για τη χρήση των ε, κανονιστικών διαδικασιών με ε, εξέταση με βάση τα άρθρα 291 και 295 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 102 τροπολογίες που υπέβαλε ο εισηγητής. Κανείς άλλος δεν έχει υποβάλει τροπολογίες. Ο εισηγητής στη Τζούρι έχει πει ότι θα περιλάβει όλες τις τροπολογίες της δικής μας Επιτροπής και των άλλων. Είναι η πρώτη φορά που η Γιούρη χρησιμοποιεί το 53-4, άρα δεν υπάρχει σχέδιο γνωμοδότηση, αλλά όλες οι τροπολογίε του εισηγητή και των άλλων υποβάλλονται ταυτόχρονα. Η πρόταση τη Επιτροπής μεταφέρει μέτρα που προηγουμένως ε, εφαρμόζονταν ε, από, μέσω της κανονιστικής διαδικασίας σε κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Και αυτό περιλαμβάνει 13 πράξεις αρμοδιότητας έκον για στατιστικά θέματα, για διεθνή λογιστικά πρότυπα, το ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες συμφωνίες. Οι περισσότερες τροπολογίες στοχεύουν να βελτιώσουν την διατύπωση του πεδίου εφαρμογή ε, και ε, θα τα προσαρμόσει στην ομολογία. Όμως οι τροπολογίες 32 και 37 αλλάζουν την ε, αντίστοιχη πρόταση από εφαρμοστική σε κατοξιδότηση. Και επίσης ορισμένες άλλες τροπολογίες αφαιρούν τη, δυνατότητα ε, ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση ανάγκης. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτά λοιπόν θέλω να πω ως Πρόεδρος. Η ΣΥΡΠΑ είναι παρούσα. Να τη δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω πως η θέση του εισηγητή είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και δεν έχω άλλες τροπολογίες ή περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν θέλει να μας πει τη γνώμη της για τις 102 αυτές τροπολογίες. Κύριε Κλάους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, μόνο 102. Αλλά να σας πω σύντομα, να αντιδράσω μάλλον σύντομα, σε κάποια σημεία που έχει εξετάσει ε, συγκεκριτή στο σχέδιο γνωμοδότησης. Εδώ η ευθυγραμμίζονται συνολικά 168 νομικές πράξεις ε, στην, ε, υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι οποίες είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Κάναμε μία προσπάθεια ευθυγράμμισης το 2013 αλλά στο Συμβούλιο δεν τα καταφέραμε γι' αυτό τώρα κάνουμε μια δεύτερη απόπειρα αλλάζοντας την νομοθετική τεχνική προτείνουμε τώρα την τροποποίηση κάθε μίας από τις βασικές νομικές πράξεις μεμονωμένα και γι' αυτό και πρέπει μαζί σας και με το Συμβούλιο να συζητήσουμε μία προς μία όλες αυτές τις τροπολογίες. Τώρα, αφού είδαμε τα πρακτικά, θα ήθελα σύντομα να αντιδράσω σε δύο-τρία σημεία Καταλαβαίνω ότι ο εισηγητής, ε, μάλλον η Κομισιόν έχει προτείνει όπως ήθιστε, μία μη καθορισμένη διάρκεια των εξοδοτήσεων. Ο εισηγητής διαρκώς, διαρκώς αλλάζει αυτό το α, επαόριστο διάρκεια στα πέντε χρόνια επί τη βάση της έκθεσης της Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει την άποψη ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Καταρχάς, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν ανα πάσα στιγμή να αναστείλουν μια εξουδότηση και έπειτα έχουμε εμπειρία. Δεν, ε, δεν ε, εισάγουμε εδώ καμία νέα ε, αξιοδότηση. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο δηλαδή. Τρίτη παρατήρηση. Με την δημιουργία αυτής της υποχρέωσης αναφοράς μετά από πέντε χρόνια για όλες τις εξοδοτήσεις, για όλους τους τομείς, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο διοικητικό φόρτο για την Κομισιόν. Κάτι ακόμα θα ξεκινήσουμε ένα νέο μητρό για τις κατεξιδότητες πράξεις στα τέλη του έτους που θα ε, μας παρέχει την πλήρη διαφάνεια για όλες τις κατεξιδότητες πράξεις σε κάθε σημείο της διαδικασίας, σε κάθε φάση μάλλον της διαδικασίας. Οπότε η διάρκεια πενταετής χρησιμοποιείται μόνο με επιλεκτικό τρόπο θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένα και με επιλεκτικό τρόπο. Επίσης, ο κύριος Γκολτιέρη επιθυμεί μία περίοδο ενστάσεων τρίμηνη συν ε, δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις μήνες. Αυτή τη στιγμή ισχύει το δύο μήνες συν δύο. Ξέρουμε ότι στον τομέα της ΕΚΟΝ, ειδικά σε κάποιες χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ισχύει το 3 συν 3 μήνες, ωστόσο δεν θα θέλαμε αυτό να ισχύσει σε, ολο, σε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να πάμε ανά περίπτωση. Υπάρχει και μια τροπολογία, πιστεύω είναι η 99, που θα ήθελα σύντομα να την αναφέρω, που η εισηγητής προτείνει να διαγραφεί η ισχύουσα εξοδότηση στην βασική πράξη, γιατί η διατύπωση δεν είναι πολύ σαφής ως έχει και ότι η εξοδότηση δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να διαγράψουμε μια εξοδότηση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμη στο μέλλον και ίσως να πρέπει να εξετάσουμε τη διατύπωση αντί να το διαγράψουμε. Δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρόμαξα μήπως μας ενημερώνατε για κάθε μία τροπολογία χωριστά. Και τώρα έχουμε το σκιώδη συγητή μας από τους πράσινους. Σας καλωσορίζω κύριε Χάουτ. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα το καλοκαίρι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για σύντομα σχόλια. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντως πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι. Περίμενα έξω μέχρι ότου να έρθει ο Πρόεδρος, αλλά δεν ήρθε. Οπότε ε, έχω προετοιμάσει ένα πολύ μακρύ, μια πολύ μακριά ομιλία για να συγχαρώ τον Πρόεδρο για τη δουλειά του. Όχι, όχι, μην τρομάζετε. Να, να συμπληρώσω μόνο αυτό που είπε η ΣΥΡΠΑ πριν από λίγο, ότι στηρίζουμε τον εισηγητή και τον πρόεδρο. Θέλουμε να τον συγχαρούμε για τη σπουδαία του δουλειά εδώ και στηρίζουμε και τι 102 τροπολογίε όσες έχουν. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να το διαβιβάσετε στον πρόεδρο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. βεβαίω και θα το, το διαβάσουμε. 100% υποστήριξη από την Επιτροπή και τις ομάδες που είναι παρούσες. Η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ ε, προβλέπεται για τις 26 Σεπτεμβρίου. Η Γιούρη δεν έχει αποφασίσει μάλλον πότε θα ψηφίσει, αλλά εμεί θα ψηφίσουμε πριν. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτω τη συνεδρίωση μέχρι τις 3. Και θα μιλήσουμε εκεί για τη CCC και τη CCCTB. Και μην ξεχνάτε, ψηφίζουμε και στις 5.